Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με την απόψινή μερίσια διάταξη έχουμε τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της οδηγίας του 2001, κάθετος 20. Θα δώσω το λόγο για 5 λεπτά στην Μισελ Ριβαζή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικός ο κανονισμός αυτός για τις ε, κλινικές μελέτες. Το 2001 υπήρχε μια οδηγία, ήδη σημαντικό βήμα αυτό για την κατάρτιση προδιαγραφών, για την εξαγωγή αυτών των δοκιμών και στην Ένωση και διεθνώς. Και κατόπιν η Επιτροπή μας είπε ότι ο αριθμός των ε, κλινικών ε, μελετών μειώνεται στην Ευρώπη και ένας από τους κύριους λόγους ήταν οι προθεσμίες και τα προβλήματα εναρμόνισης. Οπότε κοιτάξαμε εκ του σύνεγγυς ε, της διατάξης και διαπιστώνουμε τα εξής τρία. Πρώτον, πρόσβαση στα στοιχεία, διαφάνεια των στοιχείων και θα σας εξηγήσω λιγάκι περί την πρόκειται. Γιατί η δυνατότητα πρόσβασης στις εκθέσεις των ε, κλινικών μελετών και των ε, στοιχείων που έχουν συλλεγεί, με ανώνυμη μορφή βέβαια, ή η διεξαγωγή μελετών για ασθενείς σε νοσοκομεία, δηλαδή έχοντας αντικείμενο τους ασθενείς σε νοσοκομεία, είναι σημαντικό όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία για να μην ξαναγίνονται παρόμοιες μελέτες να σας ενημερώσω για κάτι που έμαθα από πρώτο χέρι. Μας ε, απευθύνθηκε σε μας ο Διευθυντής Γκίντο Ράζη της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για ένα φάρμακο που λέγεται ημιρά έδωσε έγκριση ο οργανισμός αυτός για να ε, μπει σε κυκλοφορία αυτό το φάρμακο και η φαρμακευτική εταιρεία Abbott θέλει στο site της να διαγραφούν οι κλινικές μελέτες και λένε ότι είναι θέμα εμπορικού απορρίτου και πνευματικής ιδιοκτησίας. Καλώ όλους τους συναδέλφους εδώ να υπογράψουμε μία απάντηση που θα καταρτήσουμε για να υποστηρίξουμε τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για να μπορέσει να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, δεν θέλει αυτή τη στιγμή η βιομηχανία ε, να υπάρχουν τα στοιχεία για τις κλινικές μελέτες, ενώ δόθηκε η άδεια κυκλοφορία των φαρμάκων. Επικαλούμενοι λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ ο κανονισμός μας, 1049 2001, Κοινοβούλιο Συμβούλιο, που σχετίζεται με την πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία των τριών θεσμικών οργάνων έχουμε κάθε δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση με βάση αυτόν τον κανονισμό σε αυτά τα στοιχεία. Πιστεύω ότι για όλους μας η πρόσβαση στην πληροφόρηση, τα ε, έγγραφα, τα στοιχεία, τα στοιχεία σε ακατέργαστη μορφή αλλά και στις μελέτες, φυσικά με ενώνυμη μορφή, είναι θεμελιώδους σημασίας. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο του κανονισμού αυτού, οι επιτροπές δεοντολογίας. Η πρόταση της Επιτροπής είχε σχεδόν καταργήσει αυτές τις επιτροπές. Εμείς θέλουμε την έγκριση αυτών των επιτροπών διοντολογία πριν οι εθνικέ αρχές δώσουν την έγκρισή τους για να διεξαχθούν αυτές οι κλινικές μελέτες. Γιατί η Επιτροπή Διοντολογίας ελέγχει αν έχουν ενημερωθεί σωστά οι ασθενείς, εάν τα ερευνητικά πρωτόκολλα είναι σύνομα κτλ. Θεμελιώδη λοιπόν αυτά. Τέλος, Μέσω της ε, διαφάνειας δεν θέλουμε μόνο καινοτομία, θέλουμε και προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό θέλουμε εναρμόνιση στον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών δεοντολογίας. Στην ε, Γαλλία υπάρχουν 40, στην Ιταλία 200. Και γι' αυτό μέσω των τροπολογιών μας θέλουμε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για την εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας στις διάφορες χώρες αυτών των επιτροπών για να μπορούν να διεξάγονται και μελέτες πολυεθνικές. Και κάποιους ορισμούς θέλουμε να διατηρήσουμε που υπήρχαν ε, και ήταν σωστοί στον κανονισμό του 2001 και τώρα καταργούνται με τη νέα πρόταση και θέλουμε να επανέλθουμε. Και τελευταίο θέμα. Οι κλινικές δοκιμές χαμηλής επέμβασης, χαμηλού επίπεδου επέμβασης. Ξέρετε υπάρχουν δύο επίπεδα λοιπόν. Οι κλινικές δοκιμές όπου κάνουμε πειράματα με το φάρμακο αυτό, το ελέγχουμε και μετά ένα δεύτερο επίπεδο τέτοιων κλινικών δοκιμών όπου δεν χρειάζονται ε, του ιδίου επίπεδου εγγύησης. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Ξέρετε ότι όπως είδαμε και στην περίπτωση του Mediator, που δεν χρησιμοποιήθηκε για διαβήτη αλλά για άλλα, άλλες ασθένειες. Ε, ξέρουμε λοιπόν ότι η δεύτερη αυτή μελέτη κατέδειξε κάποια ε, προβλήματα που δεν τα είχε αναδείξει η... δεν το είχαν αναδείξει οι προηγούμενες μελέτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρεμβαίνω για λογαριασμό της ε, Φρανσουάζ ε, Γκριστέτ ε, που είναι σκιώδης ηγήτρια για το ΕΛΚ. Θα ήθελα να ξεκινήσω καλωσορίζοντα την πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων Ειδικά καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν για το να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την υποβολή και αξιολόγηση των κλινικών πειραματών ανησυχώ για το ότι φεύγει η έννοια των ε, δοκιμών χαμηλής ε, παρεμβατικότητας και αυτό αφορά τις δοκιμές οι οποίες έχουν ε, χαμηλό ρίσκο. Δεν θα πρέπει εμείς λοιπόν να παρεμβαίνουμε στους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εξολόγηση των κλινικών δοκιμών. Από την άλλη, εφόσον οι επιτροπές ε, ηθικής ε, εμπλέκονται μέσω στην διαδικασία διοδότησης, θα έπρεπε να έχουμε λόγο στην ε, εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς δεν χρειάζεται ρητά να αναφερθεί κάτι τέτοιο. Επίσης η έκθεση όσον αφορά το δικαίωμα πληροφόρησης ε, για τα αποτελέσματα των δοκιμών πηγαίνει πολύ περιτέρα από αυτό το οποίο θα ήταν απαραίτητο για την ορθή πληροφόρηση και έτσι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός και οι ερευνητέ βρίσκονται σε δυσμενή θέση όσον αφορά τώρα την προστασία των δεδομένων. Η δημοσίευση θα πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες για να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες δοκιμές και για να αποφευχθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός ο οποίος ε, θα μπορούσε να απειλήσει την ευρωπαϊκή κλινική έρευνα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να δημοσιεύονται εγκαίρως και με τρόπο που θα επιτρέπει την πληροφόρηση του κοινού, των ασθενών και των ερευνητών για τα συμπεράσματα των κλινικών αυτών δοκιμών, χωρίς να εμποδίζεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Έρευνας δημοσίευση αυτών των αποτελεσμάτων είναι σημαντική για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Στην εθνική πτυχή, ο ρόλος ε, των σχετικών επιτροπών δεν φαίνεται να καθορίζεται επαρκώς ε, στην πρόταση της ε, Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία για το τι μπορεί να αναφερθεί όχι στο κείμενο σε σχέση με αυτό το θέμα. Εγώ δεν είμαι κατά τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών αυτών, αλλά δεν πρέπει να αλλάξουμε την ε, φύση του κειμένου. Τέλος, πολλές σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες ε, ασθένειες ε, δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί σωστά και δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Κλινικές δοκιμές είναι πάρα πολύ σημαντικές καθώς μπορεί να αυξηθεί η γνώση μας με την σωστή αξιολόγηση των δεδομένων. Τα δέκαρα μέλη πρέπει να γνωρίζουν αυτή την προσθέμενη αξία. Σε περίπτωση μιας σπάνιας ασθένειας, η δυσκολία σχετίζεται συχνά με τον χαμηλό αριθμό ασθενών για κάθε αρρώστια. Και βεβαίως το ότι είναι διασπαρμένη, γεωγραφικά διασπαρμένη. Σας ευχαριστώ λοιπόν, αυτά έχει να πει η Γκοστέτ. Σας ευχαριστώ κύριο Κορέα Κάμπος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας ε, τη συνάδελφο Μισελ Ριβαζή για την ε, έκθεσή της και για την ανάλυση που έκανε σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και να πω ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελματική μου ζωής που ήμουν, ε, διατέλεσα υφυπουργό ε, πολλές φορές ε, στο Υπουργείο Υγεία, δύο φορές διατέλεσα υπουργό Υγεία και εργάστηκα και ως ακαδημαϊκός ε, στην ε, ιατρική σχολή δεν είδα τέτοιες προτάσεις ε, σαν αυτές εδώ. Οι προτάσεις που γίνονται για έναν μηχανισμό ώστε να γίνει πλέον προφανές η παρακμή των κλινικών δοκιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει τρόπος, δεν Εδώ προτείνεται να γίνουν ε, τέτοιες, ε, προ... Ε, προτείνονται μάλλον τέτοιες προτάσεις που θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη παρακμή των κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη. Είναι πολύ σκληρά τα λόγια μου, αλλά ήθελα να είμαι πολύ ξεκάθαρο. Ωστόσο υπάρχουν και πλονεκτήματα σε αυτόν τον κανονισμό. Ο ορισμός ενός εναρμονισμένου σχεδίου αδειοδότησης στα κράτη-μέλη που θα επιτρέψει τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και θα επιταχύνει την ανάλυση των διαφόρων δοσιών μια νέα θηρίδα όπου θα απευθύνονται οι εταιρείε ε, αλλά και οι εθνικές αρχές, η έννοια της αξιολόγησης του κινδύνου ε, για τις κλινικές δοκιμές και η θέσπιση ενός εθνικού μηχανισμού για αποζημίωση ε, των ζημιών αλλά και για άβληση των του φόρτου, του διοικητικού αλλά και του οικονομικού όσον αφορά την προώθηση φαρμάκων. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει η παράληψη ε, όσον αφορά την διοντολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, των ασθενών. Επίσης δεν υπάρχει ενίσχυση των διατάξεων για τις ε, ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις. Όπως γνωρίζουμε, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ε, συνήθως αποσιωπούν τις, ε, τα αρνητικά πορίσματα. κάνουν τεράστιες προσπάθειες μόνο για να δημοσιεύουν θετικά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα, ενώ θα έπρεπε να δημοσιεύονται και τα αρνητικά. Ε, αποτελέσματα των δοκιμών. Ε, ανησυχούμε για το γεγονός ότι, ότι θεσπίζονται επίσης πολύ απαιτητικές προθεσμίες για την αξιολόγηση των ε, πορισμάτων των κλινικών δοκιμών. Ε, στην ουσία προωθείται μια σιωπηρή και αυτόματη έγκριση φαρμάκων. Μα αυτή δεν είναι αδειοδότηση, δεν πρόκειται για έγκριση, πρόκειται για μια μια επιστημονική διαδικασία δεν έχει να κάνει με προθεσμίες ε, και με επιβολή ε, θεσμικών προθεσμιών από πλευράς των ε, εθνικών αρχών. Θα πρέπει οι εθνικές αρμόδιες αρχές να μπορούν με πολύ μεγάλη προσοχή να εξετάσουν το κάθε ντοσιέ. Και Επίσης, το κράτος μέλος το οποίο αναφέρει ή κάνει τις ε, κλινικές δοκιμές μπορεί να οδηγήσει, ε, στη, μάλλον, το ότι επιτρέπουμε το κάθε κράτος να κάνει ε, χωριστές δοκιμές μπορεί να οδηγήσει έπειτα σε επιλογή, να μπορούμε, δηλαδή να επιλέξουμε τα αποτελέσματα που μας ε, βολεύουν κάθε φορά και η, οι έξι μέρες δε προθεσμία που δίνονται για έγκριση που πλευράς του κράτους μέλους είναι γελία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο λεπτομερής και προσεκτική ανάλυση. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, πιστεύω πως η ε, πρόθεση της Κομισιόν είναι να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική για τις κλινικές δοκιμέ και για τις έρευνες ε, της κλινική. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιδιωχθεί ει βάρος της ε, προστασίας των πολιτών των ίδιων. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ ο συνάδελφος Τζόνστον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως ε, καλώς ορίζουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν και την απλοποίηση που προκύπτει από αυτήν, γιατί έχουμε πιο εναρμονισμένες διατάξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για τις ε, κλινικές αυτές δοκιμές και σημαντικό είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία στο μέλλον η Ευρώπη θα είναι ένα σημαντικός χώρος ε, ιατρικής ε, έρευνας και για την ανάπτυξη φαρμάκων για να έχουμε καλύτερη υγειονομική φροντίδα για τους ε, συμπολίτες μας. Και νομίζω πως μια σημαντική πτυχή είναι το πώς θα έχουμε μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των συστημάτων υγείας, ανεξαρτήτως του εάν είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Η Κομισιόν πρέπει απλά να συντονίσει τα διοικητικά μεταξύ των κρατών μελών. Η πτυχή ηθική μπορεί να μείνει στο επίπεδο των κρατών μελών. Καλώς ορίζω αυτό. Και θα ήθελα να γνωρίζω επίσης ακριβώς τι στόχο έχει ο εισηγητής. Συμφωνώ όμως πως είναι σημαντικό οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες ε, δημοσίως, όπως επίσης και τα πρωτογενή δεδομένα. Αλλά σημασία έχει και η σωστή χρονική στιγμή μεταξύ δηλαδή της ε, δημόσιας πρόσβασης ε, των δεδομένων και της κυκλοφορίας του φαρμάκου. Για να δούμε και την εμπορική πτυχή και τα συμφέροντα των πολιτών. Ευχαριστώ, Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Να τονίσω τα εξής τέσσερα. Πρώτον, η σημασία των συγκριτικών κλινικών δοκιμών. Δεύτερον, το ανέφεραν ιδιαίτεροι, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση για τους πολίτες τους ίδιους. πρέπει να υπάρχει ε, ένα μητρό όπου να αναφέρονται όλα τα θέματα για την ασφάλεια για τους ίδιους τους ερευνητές αλλά και για τους αναδόχους και ένα τελευταίο που δεν έχει αναφερθεί αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πολύ σημαντικό οι κλινικές δοκιμές που γίνονται σε τρίτες χώρες, σε αναπτυσσόμενες δηλαδή Και εδώ πρέπει να ελέγξουμε τα θέματα δεοντολογίας, για τα στοιχεία, τις συνθήκες με τις οποίες συλλέγονται και την πληροφόρηση που ε, δίδεται στους συμμετέχοντες ασθενείς. Η Ένωση διεξάγει διάφορες κλινικές ε, δοκιμές σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται σεβαστές οι αρχές της δεοντολογίας αλλά πρέπει και να πληροφορούμε τους ασθενείς σε αυτές τις χώρες. Δεν γίνεται πάντα. Τονίζω τη σημασία του. Ευχαριστώ πολύ. Να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για τις τροπολογίες που προτείνει και να σας πω ποια είναι η προέλευση του θέματος αυτού. Η ισχύουσα οδηγία εκπονήθηκε για να βοηθήσει εντός εισαγωγικών τις μεγάλες, φαρμα... τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ούτω ώστε να διεξάγουν τις κλινικές τους δοκιμές σε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει ένα, ένα βαθμό εναρμόνησης αλλά 40% των ε, δοκιμών το 2007 γίνονται από ανεξάρτητους ερευνητές, από ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστημία κτλ. Και ανεξάρτητους ερευνητές. Και η εισηγήτρια αναφέρεται κυρίως σε μη εμπορικές κλινικές δοκιμές. Έχουμε πολλά στοιχεία. Όλοι οι σημαντικοί ογκολογικοί ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι θέλουν να ε, το επιτύχουμε, να επιτύχουμε με αυτήν την αναθεώρηση, να τις βοηθήσουμε. Όλες αυτές οι δοκιμές γίνονται και με βάση τις εθνικές παραδόσεις. Θέλουμε να σεβαστούμε την επικουρικότητα, δεν θέλουμε να παρέμβουμε, εφόσον όμως θα παρεμβαίνουν οι επιτροπές δεοντολογίας και γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες. Βεβαίως, ε, τέθηκαν ορισμένα θέματα. Θα τα αναφέρω όλα νομίζω. Πρώτα απ' όλα, χαμηλής παρεμβατικότητας ε, κλινικές δοκιμές είναι διεθνή και διεθνώς αποδεκτή πρακτική. Οπότε εισάγουμε αυτή την έννοια με βάση τη διεθνή πρακτική, όχι προς το συμφέρον της βιομηχανίας, του κλάδου δηλαδή. Ο κλάδος ε, κυρίως ασχολείται με την, ε, με, το, με την δημιουργία νέων φαρμάκων. Εδώ για την ογκολογία και την αιματολογία διάφοροι πανεπιστημιακοί φορείς κάνουν μελέτες για ήδη κυκλοφορούντα φάρμακα. Είπατε ως εισηγήτρια ότι δεν υπάρχει επαρκής ασφάλιση για θέματα αποζημίωσης. Υπάρχουν όμως οι κανονικοί κανόνες ευθύνη όταν παίρνετε για παράδειγμα κάποιο φάρμακο. Ισχύουν κάποιοι κανόνες, αυτοί οι ίδιοι. Γιατί εδώ χρησιμοποιούμε φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν και με βάση ακριβώς την ποσολογία και τις άλλες ενδείξεις που αναφέρονται για τη χρήση τους την δόσολογία. Ξέρετε ότι οι επιτροπές διοντολογίας έχουν διαφορετικό ρόλο στις διάφορες χώρες. Δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε επιθυμητό να υπάρξει πλήρη συναρμόνιση. Το πιο σημαντικό είναι να καθορίσουμε τις πλευρές της αποτίμησης που θα αντιμετωπίζουν από κοινού τα κράτη-μέλη ή διαφορετικά σε ομοσπονδιακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Υπογραμμίζω ότι δεν ισχύει ότι οι επιτροπές διοντολογίας δεν παίζουν ρόλο στην αποτίμηση των φαρμάκων. Έτσι γράφει στον τύπο τις τελευταίες μέρες. Αλλά επειδή έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις, είμαστε ανοιχτοί για να διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε προσεκτικά οποιασδήποτε προτάσεις και στην ένβη που είναι υπεύθυνη από τις ουσίες και στο Συμβούλιο καταλαβαίνετε ότι έχει ζητηθεί ε, διαμακρόν το θέμα. Η διαδικασία για αποτίμηση των κλινικών δοκιμών δεν θα γίνει μεμονωμένα, αλλά από κοινού από όλα τα κράτη-μέλη. Και υπογραμμίζω ότι στο τέλος της διαδικασίας οι αποφάσεις είναι καθαρά εθνικές. Η κάθε χώρα αποφασίζει αν θα εγκρίνει ή όχι κάποιο φάρμακο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απόφαση. Οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των Επιτροπών Δεντολογίας είναι εθνικές αποφάσεις. Διαφάνεια τώρα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Η διαφάνεια των στοιχείων που έχουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί και που σε, βασίζονται σε εμπορικές αποφάσεις δεν αφορά τη συζήτηση αυτού του κανονισμού, αφορά τον κανονισμό για την έγκριση κυκλοφορίας φαρμάκων. Και γενικά η διαφάνεια για όλα τα δεδομένα γενικά των κλινικών δοκιμών για οποιαδήποτε φάρμακα υπάρχοντα ή νέα. Όπως είπε η κυρία Ριβαζή, είναι θέμα του Οργανισμού Φαρμάκων. Εμείς ως Επιτροπή υποστηρίζουμε τον Οργανισμό Φαρμάκων για την ε, δημοσιοποίηση των στοιχείων μετά την χορήγηση της ε, άδεια εμπορίας. Αναφέρθηκε το χουμίρα, το φάρμακο χουμίρα. Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές. Έχει να κάνει με τον κανονισμό για την έγκριση κυκλοφορίας. Η Επιτροπή, ο Επίτροπός μου, υποστηρίζουμε σαφώς τον καθηγητή Ράζη και τον Οργανισμό Φαρμάκων στο θέμα αυτό. Θέλουμε διαφάνεια γενικά των δεδομένων της έρευνας. Το θέμα είναι τι θα είναι δημοσιεύσιμο κάποιο διάστημα, ένα χρόνο ή κάποιο άλλο διάστημα μετά το, μετά το τέλος των κλινικών δοκιμών. Θα εξετάσουμε τις προτάσεις και της κυρίας Ριβαζή και των άλλων εισηγητών στις άλλες επιτροπές. Ωστόσο, οι κανόνες που διαμορφώνουμε δεν θα εφαρμοστούν μόνο για τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και για τους μικρούς ερευνητικούς οργανισμούς. Οι εταιρείε που κάνουν αίτηση κυκλοφορία πρέπει να στείλουν στους εθνικούς οργανισμούς ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όλα τα στοιχεία και αυτοί οι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν όλα τα στοιχεία, μεμονωμένα στοιχεία, κατέργαστα στοιχεία και στην ουσία όλοι χορηγούν αυτά τα στοιχεία με πολύ ε, μικρό ποσοστό ε, εμπιστευτικών στοιχείων που δεν δημοσιεύονται για λόγους εμπορικούς όπως για παράδειγμα τη διαδικασία παραγωγής. Βεβαίως, όταν λοιπόν ζητηθεί η έγκριση κυκλοφορίας, χορηγούνται όλα αυτά τα στοιχεία. Παρακαλώ, ρωτήστε και τους ερευνητές, ρωτήστε τους πανεπιστημιακούς, θα διαπιστώσετε ότι οι κλινικές δοκιμές που γίνονται για σοβαρά φάρμακα μπορούν να σώσουν ζωές, Ρωτήστε τους αν είναι σε θέση να ε, εκπληρώσουν αυτές τις ε, υποχρεώσεις εάν δεν έχουν στόχο να αιτηθούν κυκλοφορία φαρμάκου. Λόγω της ε, προθυμίας με την οποία έχουν ασχοληθεί διάφορες επιτροπές του σώματός σας με το θέμα αυτό, ελπίζουμε ο κανονισμός αυτός να εγκριθεί πριν το τέλος της τρέχουσας θητείας. Διότι η οδηγία αυτή δημιουργεί δυσχέρειες για τις μη εμπορικές δοκιμές και τους μη εμπορικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Δημιουργεί λοιπόν δυσχέρειες αυτός ο υπάρχον κανονισμός και πρέπει να αναθεωρηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η Μισελ Ριβάζη. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους τους και τους κοιόδης εισηγητές για αυτή την γνωμοδότηση. Εγώ πιστεύω πως συμφωνούμε περίπου όλοι για την προστασία των ασθενών, για την Επιτροπή Ιδιοντολογίας, για τα στοιχεία κτλ. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο γίνεται μια συνάντηση με την παρουσία της Κομισιόν καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Πρέσκρε που είναι μια ένωση ανεξάρτητων γιατρών για να εξετάσουμε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της πρόσβασης στα στοιχεία και των βάσεων, στις βάσεις δεδομένων. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία. Ο ένας είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο δεύτερος η Κομισιόν. Πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να το ανορμανίσουμε γιατί ο οργανισμός είναι η έγκριση για εμπορία φαρμάκων, ε, η Κομισιόν ε, είναι η έγκριση για τις ε, μελέτες των ερευνητών, αλλά διαρωτώ μου πως όλα αυτά πρέπει να τα ενώσουμε σε μια κοινή βάση. Η αυρενή συζήτηση λοιπόν σε αυτό θα ε, ε, μας απασχολήσει και ε, θα τα πούμε αύριο λοιπόν για μια συνεδρίαση από αυτές τις βάσεις. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ. Η... 26 Φεβρουαρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών το μεσημέρι στις 12. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά το άρθρο 70 παράγραφος 4 του κανονισμού επί τη βάση του οποίου καλούμεθα να ενημερώσουμε για τις εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Θα ξεκινήσω δίνοντας τον λόγο, επειδή δεν είναι όλοι στην αίθουσα, στον συνάδελφο Μπέλετ. Είναι παρόν, από ό,τι μου είπαν. Παρακαλώ για την κατάσταση πρόοδου όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους που έχουν γίνει και αυτόν που θα γίνει αύριο. Παρακαλώ. Τρία λεπτά έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, γιατί έχουμε τις ψηφοφορίες στις 4. Θα σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση πρόοδου Έχουμε και τον ε, τριμερή διάλογο που γίνεται αύριο το πρωί. Νομίζω πως έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της αυριανής συνεδρίασης, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε σε τελική συμφωνία για συμβιβαστική. Να πω κάτι αρχικά για την εμπτουσία αυτής της πρότασης οδηγίας. που είναι η απόλυτη ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια την ασφάλεια των εργαζομένων στις ε, πλατφόρμες εξόριξης ε, στην ανοιχτή θάλασσα και από την άλλη πλευρά η εγγύηση για τον ε, έλεγχο του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και φυσικά ε, το Κοινοβούλιο είναι υπέρ ε, ενός συνικού τείχους όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών πτυχών και των αρχών εντός του Εθνικού Διοικητικού Μηχανισμού που είναι υπεύθυνε για το οικονομικό στοιχείο, για τα έσοδα δηλαδή τέτοιων επιχειρήσεων ανοιχτής θάλασσας. Είμαστε στο δρόμο για μια καλή συμβιβαστική ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το σημαντικό στοιχείο αυτής της νέας οδηγίας. Ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό είναι το θέμα των ευθυνών. Ποιος δηλαδή είναι κάθε φορά υπόλογος. Ποιος φέρει τις ευθύνες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, για τα οικονομικά ζητήματα, σε σχέση με τις επιχειρήσεις ε, ανοιχτής θάλασσας και το Κοινοβούλιο έχει καταφέρει να πετύχει το στόχο του εδώ πιστεύω γιατί βέβαια είπαμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές ευθύνες, δηλαδή οι φορείς που λειτουργούν offshore θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα την τεχνική αλλά και την οικονομική για να καλύψουν οποιασδήποτε πιθανές περιβαλλοντικές ή οικονομικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τις ε, δραστηριότητές τους. Και έχουμε φτάσει σε συμφωνία για αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα προσφυλές για στο Κοινοβούλιο, είναι φυσικά η πτυχή της συμμετοχής ε, του ε, δημοσίου, δηλαδή σε όλες τις φάσεις τέτοιων δραστηριοτήτων, ε, έρευνα, παραγωγή, το κοινό να μπορεί να ενημερώνεται. και σε αυτό το σημείο πιστεύω πως αύριο το πρωί θα βρούμε συμφωνία γιατί είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι η ενημέρωση του κοινού θα είναι κομμάτι αυτής της νέας οδηγίας. Νομίζω πως είναι ήδη και εκτιμένο. Δεν το έχουμε πετύχει 100% αλλά κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, μια τελευταία παρατήρηση, κυρία Σαρτόρη, αφορά την ε, παγκόσμια διάσταση, γιατί είναι ακόμα αυτό ένα στοιχείο το οποίο έθεσε το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, η ε, παγκόσμια απόδοση των ευρωπαϊκών εταιριών πρόκειται για μια οδηγία που ισχύει για την επικράτεια και τα ύδατα της Ένωσης και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά τις εταιρείε μας. Οι εταιρείε όμως που δραστηριοποιούνται εντός των ευρωπαϊκών υδάτων υποχρεούνται να αναφέρουν αντιστοιχήματα εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων στις αρχές της Ένωσης. Συνοψίζω δηλαδή ευρωπαϊκές εταιρείες ή μάλλον εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες, καταχωρημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δραστηριοποιούνται και εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβεί κάποιο δυστύχημα υποχρεούνται να αναφέρουν το εν λόγω δυστύχημα στις αρχές της Ένωσης έτσι ώστε να μπορούμε να αποκομίζουμε τα διδάγματα από αυτά τα δυστυχήματα. Ένα δεύτερο στοιχείο που αφορά την παγκόσμια διάσταση αυτής της οδηγίας είναι ότι η πολιτική πρόληψης Δηλαδή το έγγραφο, όπως ονομάζεται, πολιτικής πρόληψης μεγάλων ε, δυστυχημάτων, ε, θα πρέπει να ε, ισχύει μόνο για τέτοιου είδους δραστηριότητες εντός των υδάτων της Ένωσης, αλλά και εκτός των υδάτων της Ένωσης. Γιατί διαπιστώσαμε ότι το στοιχείο της πρόληψης θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις δραστηριότητες των ε, εταιριών που είναι γεγραμμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία παρατήρηση ε, αφορά την Αρκτική. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις και τροπολογίες που κατητέθησαν από απαγόρευση, μορατόριο για εξόρυξη στην Αρκτική μέχρι την ε, τροπολογία που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου Φυσικά δεν θα υπάρξει απαγόρευση ε, δραστηριοτήτων στα νυχτά στην Αρκτική για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά ύδατα στην Αρκτική. Άρα οι νομικές μας αρμοδιότητες είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με αυτό το θέμα. Ωστόσο, εταιρείε που θα είχαν την πρόθεση να, ευρωπαϊκές εταιρείες που θα είχαν την πρόθεση να αρχίσουν δραστηριότητες offshore στα ύδατα της Αρκτικής, θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό, αυτό μπορέσαμε να το βάλουμε μέσα, δηλαδή την ε, δυνατότητα ανταπόκρισης και αντίδρασης σε πετρολοκυλίδες. Πρέπει δηλαδή κάθε εταιρεία να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να αντιμετωπίσει πετρελοκυλίδες σε πολύ δύσκολες ε, καιρικέ ή περιβαλλοντικές συνθήκες. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αποδείξει η εταιρεία ότι σε περίπτωση τέτοιες δυστυχήματος σε τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες θα μπορούσε να είναι ερκτική αλλά μπορούν να είναι και δύσκολα σημεία της Βόρειας Θάλασσας, της Μεσογείου. Θα μπορούσε αυτό να γίνει οπουδήποτε όταν μιλάμε για δύσκολε περιβαλλοντικές ή καιρικές συνθήκες. Ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι ότι οι δραστηριότητε θα πρέπει να περιοριστούν ή και να πάψουν. Έχουμε λοιπόν μια καλή εγγύηση ότι ο αντίκτυπος πιθανού δυστυχήματος θα περιοριστεί όσο γίνεται ε, περισσότερο. Αυτή είναι η κατάσταση πρόοδου πρόεδρε. Συνεχίζουμε φυσικά τις επαφές με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς απόψε και αύριο το πρωί. Ελπίζουμε πως θα έχουμε υπό την Προεδρία σας έναν πολύ αποδοτικό τριμερή διάλογο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μπέλετ που λόγω του πάυσος για αυτό το θέμα μας κρατήσατε για 7,5 λεπτά. Την επόμενη φορά θα φροντίσουμε να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο για να μας ενημερώσετε και τώρα θα δώσω το λόγο στον και συνάδελφο Μαρινέσκου ζητώντας του να κάνει πιο γρήγορα για να μας μιλήσει πιο σύντομα για το Γαλιλαίο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ξεκίνησα τις συζητήσεις με την ε, Ιρλανδική Προεδρία τελείως διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη Προεδρία. Σε δύο συναντήσεις ε, διατρέξαμε όλο το κείμενο. Σε δύο πράγματα μόνο δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Το ένα αφορά, όπως φαντάζεστε, τις ε, πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση, που θα το συζητήσουμε τελευταίο, και το άλλο σχετίζεται με την πρόταση του Κοινοβουλίου για τις ε, αιτήσει. Νομίζω πως ε, το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό θα καταλήξει σε μια πρόταση για το τι θα γίνει με τα κονδύλια του Γαλιλαίου. Αυτά και μετά θα έχουμε και μια τεχνική συνάντηση, θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και μπορούμε να προτείνουμε κάποια αποτελέσματα του τριμερού διαλόγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το συνάδελφο Μαρινέσκου για την ε, συντομία του. Τώρα, αλλά θα είναι σύντομο βέβαια γιατί έχει γίνει μόνο μία συνάντηση. Άννα Μαντουρέλ και Καρβάγιο. Να μας πούνε σύντομα την κατάσταση του τριλόγου για το ορίζον. Παρακαλώ. Ριέρα Μαδουρέλ πρώτα. Πολύ σύντομα. Άπειτη συνάδελφη. Ο κανονισμός για το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζοντας 2020 ε, είναι αντικείμενο τριμερούς διαλόγου που έχει προχωρήσει αλλά ανησυχούμε διότι οι πρόσφατες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορούν να επηρεάσουν αυτή την πρόοδο που έχουμε επιτύχει. Και μιλάω μόνο για τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Κάθε εβδομάδα έχουμε τεχνικές συναντήσεις, όπου μέχρι στιγμής έχουν ζητηθεί τα άρθρα του κανονισμού. Ίσως αυτή την Παρασκευή θα μπορούσαμε να έχουμε μια ε, αρχή συμφωνία για το σύνολο των άρθρων. Το Κοινοβούλιο παίζει ε, σκληρό παιχνίδι, προσπαθεί να διατηρήσει τα στοιχεία κλειδιά, για παράδειγμα πρόσβαση, το θέμα του φύλου και η μη διάκριση, η έλλειψη διακρίσεων. Αυτά τα θέματα τα συζητάμε και σε πολιτικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως είπε και η Πρόεδρος, έχουν γίνει δύο τριμερείς διάλογοι για το θέμα αυτό. Ο πρώτος για να γνωριστούμε και το δεύτερο για να συζητήσουμε σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Συζητήσαμε και για τη δομή του προγράμματος και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο προτείνει δύο σημαντικά θέματα. Διεύρυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο και υπεύθυνη επιστήμη. Μετά μια πρώτη προσέγγιση για τα θέματα αυτά μπορώ να σας πω ότι επί του περιεχομένου θέση μας είναι κοντά στη θέση του Συμβουλίου. Αλλά δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία για το πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε το πρόγραμμα, διότι εμείς θέλουμε να υπάρχει χωριστός προϋπολογισμός και διαφοροποιημένος για τους δύο βασικούς στόχους. Για το θέμα του προπολογισμού, όπως είπα, έχουμε μεγάλη ανησυχία. Η πρόταση του Συμβουλίου είναι απαράδεκτη. Εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από τις διακηρύξεις από τη μία για επενδύσεις ε, στην καινοτομία και την έρευνα και το δημοσιονομικό πλαίσιο από την άλλη που από ό,τι φαίνεται θα μειώσει τον προπολογισμό του 2020, του ορίζοντας 2020 κάτω από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν πάμε κάτω από το 80 δις που είχαν αρχικά προταθεί στέλνουμε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα που θα μειώσει την αξιοπιστία της Ένωσης και τη δυνατότητά μας στο μέλλον να έχουμε ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Στο τέλος, οποιαδήποτε τελική συμφωνία για το πρόγραμμα Horizon 2020 εξαρτάται από επαρκή χρηματοδότηση. Εμείς ως Επιτροπή έχουμε ζητήσει φιλόδοξο προπολογισμό. Αυτός θα πρέπει να είναι και στο μέλλον ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Όσο θα προχωρήσουν οι τριμερείς διάλογοι, θα συνεχίσουμε να σας πληροφορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καρβάλιο. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, τον εισηγητή και τους και το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την καλή συνεργασία. Ιδιαίτερα καλωσορίζω το πνεύμα της Ιρλανδικής Προεδρία που είναι διατεθειμένη να συζητήσει τον ορίζοντα 2020 σε ένα πακέτο και να ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα θύματα τα οποία σύμφωνα με τον εισηγητή αποτελούν μέρο του. Όπως είπε και η κυρία Ραμαδουρέλ, είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις. Η πρώτη ήταν μια αναρακτήρια, η δεύτερη είχε περισσότερο χαρακτήρα εργασία και κυρίω είδαμε ποια είναι τα βασικά σημεία που είναι ακόμα ανοιχτά, στα οποία διαφέρομαι και είναι σημαντικά και θα έλεγα πως ε, αφορούν την διεύρυνση της συμμετοχής, της συμμετοχής, τις συνέργειες ε, των ε, διαφόρων κονδυλίων, τον ορισμό των επιστημονικών πάνελ, στον καθορισμό των πραστηριοτήτων και επίσης την δομή και το πώς μπορεί να επηρεάσει η γενικότερη επιστημονική έρευνα την ε, κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν κάποια έγγραφα τα οποία έχουν πάει από την Προεδρία, στην Προεδρία με και εξηγούν την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά τα ζητήματα. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω αυτό το οποίο είπε η κυρία Ριέρα Μαδουρέλ Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα του Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα έπρεπε να έχουμε υψηλότερο προϋπολογισμό και θα παρακολουθούμε από κοντά τις διαπραγματεύσεις ε, του Πουδοπού. Και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε υψηλότερο προϋπολογισμό, να έχουμε ένα ισχυρό πρόγραμμα το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη για την ανάπτυξη και τις δουλειές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να τονίσουμε την συνένεση που έχουν όλες οι ομάδες ε, στο ζήτημα του ότι θα είναι μοιραίες οι προτινόμενες ε, περικοπές των πυρώνα 1α ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Πρέπει να πούμε πως ε, το Συμβούλιο έχει ε, εδώ πέρα υπονομεύσει τους δικούς του στόχους για το 2020 και πρέπει όλοι μαζί από κοινού να μην αποδεχτούμε αυτόν τον προπολογισμό. Τώρα, είχαμε την πρώτη επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων ανταλλάξαμε τις βασικές μας απόψεις, δηλαδή την ε, διοικητική απλούστευση και τη μείωση του χρόνου εκταμίευσης, ε, στο οποίο συμφωνούν όλα τα θεσμικά όργανα. Οι διαφορές είναι στο πώς θα τα επιτύχουμε και βεβαίως ε, πώς θα προσανατολιστούμε στις απαιτήσει των ενδιαφερομένων. Εμείς λοιπόν θεωρούμε πώς εκπροσωπούμε και την ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και αυτό το οποίο ζητάνε. Δηλαδή να διατηρηθεί ως εναλλακτική χρηματοδότηση του πλήρους ε, κόστους, μια διαδικασία γρήγορη, γρηγορότερη εκταμίευση και θεωρώ πως πρέπει να προχωρήσουμε τώρα σε εντατικές ε, συζητήσεις και αυτά τα οποία έχουμε εμείς ως βασικές θέσεις είναι οι κοινέ θέσεις ε, όλων των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 και στο μελλοντικό ορίζοντα 2020, τα οποία είναι και τα πανεπιστήμια και η βιομηχανία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και η ερευνητική κοινότητα γενικώ. Και ως εκπρόσωποι λοιπόν όλων αυτών θεωρώ πως είμαστε σε μια καλή διαπραγματευτική θέση. Ωραία, σας ευχαριστώ. Σε τρία λεπτά θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Είχαμε ακόμα εκείνη το τριμερή διάλογο για του συναδέλφου Κρέασμαν. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο χρόνο, το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Αν ε, θέλετε, μπορείτε και τώρα να το παρουσιάσετε στα γρήγορα, αλλά καλύτερα την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, ευχαριστώ. Bene, allora possiamo... Ωραία, λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δώσαμε την άδεια να είναι παρούσα εδώ μια τηλεοπτική ομάδα, όπως είδατε. Ε, un primo voto. Και έτσι περνάμε στη πρώτη ε, ψηφοφορία, μια δοκιμή να κάνουμε. Να δούμε αν λειτουργούν ε, όλα τα μηχανήματα. Παρακαλώ, ψηφίστε. Testing vote. Check. Ωραία. Ψι... Έχετε βάλει 43 κάρτε. μόνο 37 ψήφισαν. Περνάμε λοιπόν στην ισοφορία της έκθεσης Τσίτσεστερ. Παρακαλώ κύριε Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε επικείς μαζί μου γιατί θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για το περιεχόμενο του Οργανισμού της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών ΕΝΗΣΑ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία και επίσης τα μέλη της ε, γραμματείας μας, ιδιαίτερα τον Πίτερ Τράιλ, που δούλεψε σκληρά. Χρειάστηκε να συνεργαστούμε με μια σειρά από διαδοχικές προεδρίες και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ιρλανδική Προεδρία όπου καταλήξαμε, αλλά και οι προηγούμενες τέσσερις-πέντε. ήταν η εταίροι σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Ελπίζω να είναι καλό το αποτέλεσμα. Ζητώ συγγνώμη που είναι τόσο περίπλοκη η ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά ελπίζω ότι θα τα βγάλουμε πέρα και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κύριε Τσίτσεστερ. Οπότε ψηφίζουμε το συμβιβαστικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα κάνουμε δύο ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Ωραία. 47 υπέρ, 1 κατά. Καμιά αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, συνάδελφε Τσίτσεστερ. Και ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Τέλος της ψηφοφορίας. 48 υπέρ, 2 κατά, καμιά αποχή. Έγκρινεται. Ε, Περνάμε στην έκθεση του συναδέλφου Σον Κέλλη. E Είναι κάπως πολλές οι τροπολογίες, οπότε υπομονή. Τροπολογία 304, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 305. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε για την 305 Ρούμπεκ. Ένας πράσινος παραπάνω ψηφίζει. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ, κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για 306. Τέλος της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 26 κατά. Αντιστράφηκε. Γιατί λέτε όχι. Παρακαλώ πείτε μου τι στρέχει. Με το μικρόφωνο. Ναι, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, αλλά οι δικές μας ψήφοι δεν την υπόψη γιατί δεν λειτουργήσαν το, τα μηχανήματα και είμαστε υπέρ και οι δυο μας. Ήσασταν υπέρ ή κατά. Υπέρ. Και οι δυο. Ψηφίσατε αλλά δεν λειτουργήσε το μηχάνημα. Να, κοιτάξτε. Ας κάνουμε άλλον έναν έλεγχο. Ας ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε. Voto Τέλος της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 307. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 310. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες από κοινού 21, 311, 312 και 313. Υπέρ. Κατά. υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 317 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 320 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 320 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Anche più Τέλος 21 υπέρ, 36 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 321 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 323. Α, θέλετε να ελέγξουμε τη συμβαστική. Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβιβαστική 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Κιούζα. Τέλος της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, εγκρίνεται, διορθώνει η πρόεδρος. 323. Εδώ μου λένε ότι την 323 πρέπει να την ψηφίσουμε ως προσθήκη. Τι λέτε κύριε Σιγητά Κέλλη. Ναι, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 323. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 329. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 332. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, από κοινού, 334, 335 και 336. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ και 20 κατά. 337 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέρτα. Έλεγχος ηλεκτρονικός, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος πληροφορία. 37 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. 342 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός για 342. Τέλος ψηφοφορίας. 15 υπέρ 44 κατά. Απόρριπτεται. Τροπολογία 343. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 341. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 346 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα από κοινού Ζητώ συγγνώμη, δεν παρακολούθησα. Τι έγινε με την 353. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, πήγατε λίγο γρήγορα εκεί και το έχασα. 355 δεν ψηφίζουμε. 354 την ψηφίσαμε και απορρίφθηκε. Και τώρα πάμε Στην επόμενη σελίδα, τροπολογίες 27 και 356 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Αχ, όχι, έκανα λάθος, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, ας ελέγξουμε για την 28 και την 356. Κιούζα. τη ψηφοφορία. 37 υπέρ 21 κατά. Τροπολογία λοιπόν. Εγκρίθηκε λοιπόν. 3.57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 361 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέξουμε τη συμβαστική 38. Παρακαλώ. Πέρας, 37 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 364 υπέρ. 364 υπέρ. 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40. Παρακαλώ. Ωραία, να ελέγξουμε την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 35 υπέρ 24 κατά. «25 κατά λοιπόν, ωραία. 35 υπέρ 25 κατά. Εγώ πάντα αποδέχομαι τις ε, αιτήσει για έλεγχο, ακόμη και ένας άνθρωπος να το ζητήσει, αλλά, αλλά ε, δείξτε μου κάποια εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Συμβαστική 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 373 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική, συγγνώμη, τροπολογία 375 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 375. Votazione 40 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 3,78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3,79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3,82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 384 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Από κοινού 387 και 388 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία να αλλάξουμε 32. Άρχεται η ψηφοφορία. ancora 36 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 33. 389 και 390 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 391. Υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί 35 και 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 3.96 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτονται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά αποχές. Α, να ελέγξουμε. Καλά, να ελέγξουμε. 43. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω ψηφίζει. Ωραία, εντάξει. Πέρας. 49 υπέρ, 40 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 400 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 402 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 404 υπέρ πώς 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού 40 και 406 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 408 υπέρ «408 λέω, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 44, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 412 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 419 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 424 υπέρ. 424 4.24. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από κοινού. 45 και 4.25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 4.26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 427 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 434 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 435 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 436 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 438 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.40 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 4.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού 46 και 4.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 4-4-4 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε να ελέγξουμε την 4-4-4 Πέρας. Allora, respinto. Απορρίπτεται. 4.43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4.45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 4.51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 456 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 458 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 464 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 465 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 468 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 469 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 478 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού 479 και 480 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 483 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 487 υπέρ κατά αποχές Μ, ας ελέγξουμε άρχεται Πέρας. 11 υπέρ 48 κατά. Με συγχωρείτε δεν είδα καλά. Απορρίπτεται. 4-8-7 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4-88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4-89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από κοινού. 60 και 4,90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 4, συγγνώμη, συμβαστική 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4,97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4,99 υπέρ Κατά. Ωραία, καταπίπτει το 498. Οπότε περνάμε στην 499 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 500 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 501 και 502. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 508 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 508 παρακαλώ. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 43 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 509 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 510 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 511 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 515 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 518 υπέρ Ένα λεπτό παρακαλώ. Να Σταματάμε ένα λεπτό. Πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία 69. Την βρήκατε. Μετά από την συμβιβαστική 59 που έχει αποσυρθεί υπάρχει τροπολογία 69 Πρέπει να την ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 69, παρακαλώ. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 518 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 519 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 521 υπέρ. Κατά. Όχι, 20 έχει καταπέσει. Περνάμε στην 521. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 527. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 528 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 529 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 530 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 531 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είναι ταυτόσημες οι 532 και 533. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 534 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί 534. Πέρας πληροφορίες 24 υπέρ 34 κατά. Απορρίπτεται. 535. 535. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 536. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 537. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 532 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 541 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 543 και 44 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 547 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 547. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού 548 και 549 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 551 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 552 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 553 και 54 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 73. 557, 558 και 559 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρινώνται. 561 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 562 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 563 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 564 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 565 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 566 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 567 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 568 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 569 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 570 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 571 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 572 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 573 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 574 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 575 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 576 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 577 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 578 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 579 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 580 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 583 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 584 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 585 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 586 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 587 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 588 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 77 και 589 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 78 υπέρ κατά αποχές δεν είδα καλά. 78 ας ξαναψηφίσουμε υπέρ ποιοι είναι. 78 Α, ηλεκτρονικός έλεγχος εντάξει. 31 υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 593 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5, 6, 7 υπέρ. Όχι, εγώ το είδα. Έκανα λάθος. Εννοούσα 597, όχι 567. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 602 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από κοινού, 79 και 603 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 604 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 605 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 605. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ναι. ναι, non votiamo perché è decaduto. Έχει καταπέσει. Να Δεν, χρειά... Δεν το ψηφίζουμε. 605 λοιπόν έχει καταπέσει. 80 και 606 από κοινού υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 609 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 611 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 611. Bene, votazione chiusa. Τέλος της ε, ψηφοφορίας. Λοιπόν, 8 υπέρ, 48 κατά, απορρίπτεται 611, 612 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 621 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 622 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 623 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Από κοινού 624, 625 και 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 633 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 635 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται από κοινού 636 και 637 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται από κοινού 638, 639 και 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 645 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 646 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 654 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 655 και 56 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίν, ε, απορρίπτονται. 657 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 658 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Από κοινού 85, 659 και 660 υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 662 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 663 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 664 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 665 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 666 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 667 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 668 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 69 Πέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 671 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 672 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού οι 673 και 675 υπέρ κατά από... Α, έχουν καταπέσει. Δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε. Πάμε λοιπόν στην 677 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 678 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 679 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 680 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 681 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 685 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 689 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 690 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 700 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 702 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε απορρίπτεται, με συγχωρείτε. 703 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 73, ε, 706 και 707 από κενό. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 709 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 710 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 711 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 713 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 715 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 και 716 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 76 υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Compromesso 76. Συμβαστική 76. Votazione aperta, votazione chiusa. 32. Τέλος ψηφοφορίας 32 υπέρ 27 κατά Τα 7-23 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 724 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 725 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 728 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 729 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 734 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 735 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 736 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 737 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 738 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 739 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 740 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 741 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 742 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 744 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 747 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 751 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 752 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 753 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 754 υπέρ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 764 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 765 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 766 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 767 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 768 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 769 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 770 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 771 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 773 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 777 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 778 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 780 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 781 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 782 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 783 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 784 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 787 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 788 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 789 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 791 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 792 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 793 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 794 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 795 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 796 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 797 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 798 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Από κοινού. 799 και 112 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται. 800 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 801 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 83 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 803 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 704 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 806 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 807 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 808 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 809 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού 810 και 811 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 813 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 814 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 815 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές 816 υπέρ κατά αποχές 817 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 818 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 819 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 820 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 821 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβαση 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 8.26 και 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8.28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8.29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 846 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 847 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 848 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται. 849 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 852 υπέρ κατά αποχές 51 ε, με υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 852 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 853 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 856 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 855 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 857 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 86. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 864, 863, 865 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 808 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο, συμβαστική 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 871 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 872 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 879 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 880 και 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 882 και 883 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 884 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 και 885 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 886 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 887 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού οι 157 και οι 888 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 897 υπέρ 895 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 896 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 897 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 898 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 899 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 900 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 901 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται. 902 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 903 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 904 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 905 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 906 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 908. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από κοινού 909 και 910 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 912 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 914 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 916 Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Συμβιβαστική 90, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 916, καταπίπτει και περνάμε στην 917. 917 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165, 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τι θέλετε, το 168 να ελέγξουμε. Μάλιστα, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 168 aperta. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 28 a 29 contro. 28 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Εκατόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180... Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 183. Έχετε δίκιο, είχε εγκριθεί. Ναι, εγώ έκανα λάθος, τι είπα. Τέλος της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 18 κατά. Ναι. Είδα σωστά, αλλά είπα λάθος. Ε, ήμασταν στην 183. Τώρα πάμε στην 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 και 197 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική 10 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 10. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. 27 υπέρ 32 κατά. Η συμβιβαστική 10 απορρίπτεται. Περνάμε στη 211 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Prego. 211 No, dobbiamo votare prima il 211 e il 212 perché il compromesso Πρέπει να ψηφίσουμε τη 211 και 12 γιατί η συμβαστική 10 απορρίφθηκε. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε για τη 211 και τη 212. 212 e λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 213. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 214. Υπέρ. Κατά. Τροπολογίες απορρίπτεται. 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 και 17 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, τροπολογία 226. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Υπέρ Τη συμβαστική 14 κατά αποχές εγκρίνεται. 229. Τροπολογία 229 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται, συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200, ε, συγγνώμη, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 234 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 252, 53 και 54 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 255 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 263. Υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 15 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά υπέρ, ε, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 277 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 278 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά 284 γιατί έχει καταπέσει η συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 287 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 288 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 294 και 295 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 297 ε, γιατί είχε καταπέσει η συμβαστική. 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 298 29, ε, συμβαστική 29, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 303, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, παρακαλώ. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 24. 33 υπέρ 24 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και ευχαριστώ όλους σας για την υπομονή και για την ψηφοφορία. Κυρία Τικάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ το προσωπικό των πολιτικών ομάδων για τη δουλειά που έχει κάνει. Είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις. Θα ήθελα να τονίσω δυστυχώς πως ο τρόπος με τον οποίο εργαστήκαμε δεν ήταν ο καταλληλότερος. Ο κατάλογος των ψηφοφοριών άλλαξε το βράδυ. Κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες αποσύρθηκαν και είδα πως ε, παρά το ότι κάποιες ε, πολιτικές ομάδες συνυπέγραψαν συμβαστικές προτάσεις, σήμερα τις καταψήφισαν. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες τροπολογίες. Κάποιες άλλες αποσύρθηκαν κτλ. Θα ήθελα να πω λοιπόν πως ίσως η μέθοδος εργασίας δεν ήταν η καταλληλότερη και ελπίζω στο μέλλον, ε, κυρία Πρόεδρε, μαζί με τους συντονιστές, θα ορίσετε ένα χρονικό όριο για το μέχρι πότε μπορούν να γίνονται αλλαγές ε, στον κατάλογο των ψηφοφορίων. Παρ' όλα αυτά, ε, ευχαριστώ όσους εργάστηκαν για τον κατάλογο. Ευχαριστώ, κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για την ενεργητικότητα και την υπομονή τους για πάνω από χίλιες ε, ψηφοφορίες που κάναμε και για το ότι παρέμειναν συγκεντρωμένοι και ευχαριστώ και εσάς κυρία Πρόεδρε για την αποτελεσματική διεξαγωγή της ε, ψηφοφορίας και την Πιλάρ και τον Τομπίας την συντονιστριά μας και τον σύμβουλό μας και όλους όσους ε, συνέταξαν σε αυτές τις ε, τροπολογίες ε, πάρα πολύ γρήγορα. Εξάλλου, εμείς είμαστε η βασική και κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή, οπότε έπρεπε να εργαστούμε την πράσινη εβδομάδα. Είχαμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, κάποιες αποσύρθηκαν, δικαίωμά τους ήταν. Οι ε, χρονικοί περιορισμοί λοιπόν ήταν δύσκολοι, αλλά ταυτόχρονα είχαμε πολλές ε, συζητήσεις, εργάστηκαν πάρα πολύ ισχυώδεις, ε, τους ευχαριστώ και τώρα έχουμε μια ξεκάθαρη θέση από την Επιτροπή μας προς το μέλλον. Αυτό χρειαζόμασταν. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Εγώ και κάποιοι άλλοι βεβαίω έχουμε την πόρτα μας ανοιχτή, ακούω τους πάντες, είχα γύρω στις 200 συναντήσεις ε, δέχτηκα κάποια πράγματα και οπωσδήποτε δεν με επηρέασε κανείς υπερβολικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αν θεωρούσα πως κάτι ήταν σημαντικό, το συμπεριέλαβα. Αυτό ισχύει για μεγάλες εταιρείες, ε, μικρομεσαίες, ε, ΜΚΟ, ευρωβουλευτές, το προσωπικό της Κομισιόν κτλ. Ήταν λοιπόν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, ήταν τιμή μου και βεβαίω ε, έγινε νομίζω και με πάρα πολύ μεγάλη εργατικότητα και με κάποιο έτσι πνεύμα που επιδείξαμε. Ευχαριστώ. Και αν ε, θέλετε ελάτε να πιούμε μια γκίνες πριν αρχίσει η Σαρακοστή. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω πως η επόμενη συνεδρίαση είναι 18 Μαρτίου το απόγευμα και 19 όλη μέρα. Να σας θυμίσω επίσης ότι θα γίνει ένα σεμινάριο την 5η 21 Φεβρουαρίου από τις 3 με 8 υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες. Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν. Ευχαριστώ.